επιβατικά και εμπορικά οχήματα. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Γιάβο έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο. Yes, please. Please. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ήθελα να παρουσιάσω αυτή την ένσταση όσον αφορά το άρθρο 106, όσον αφορά τα οχήματα αυτά, όσον αφορά το Euro 6, Euro 6 η ρήπανση αυτή ε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χάνονται σαν αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής κατάστασης. Ιδιαίτερα τα οξύδια του αζότου είναι κύριοι ρηπαντές και δημιουργούν καρκίνο του πνεύματος και πολλές ε, ε, αναπνευστικές ασθένειες και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και το θέμα της ε, οξύτητας ε, του ατμοσφαιρικού αέρα που είναι ε, επιβλαβή στην υγεία. Και έχουμε πολλά ε, θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσια. Βλέπουμε ότι τα, οι εκπομπές ρήπων από το diesel, τα οχήματα diesel επιβαρύνουν το περιβάλλον και η έχουμε 80 ε, χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το ε, σχέδιο που στοχεύει στο να δημιουργήσει τις πραγματικές τιμές που θα απαιτούνται από πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα. η πρόταση ψηφίσματος εξετάζει ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα οδηγούσε σε μια μια εξαίρεση εφαρμογής των ε, οριακών τιμών, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με τον στόχο που έχουμε ε, για το, από το 2007 και ξεπερνά τις αρμοδιότητες εφαρμογής σε σχέση ε, με τις διατάξεις του 2005. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει λοιπόν ένσταση εδώ την οποία υποβάλλει όσον αφορά τα οχήματα αυτά για την εκπομπή 160 ε, ε, ε, των σωματιδίων του οξυδίου του αζότου και πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη σε σχέση με το 2019. Τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά από την έναρξη σε ισχύ του, της διάταξης για το Euro 6, το Euro 6, την κατηγορία αυτή. Και υπονομεύει όχι μόνο η κατάσταση αυτή τον ίδιο τον κανονισμό, αλλά και την ίδια την αξιοπιστία της ρυθμιστικής αρχής στην Ευρώπη. Γι' αυτό το ψήφισμα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού αυτό και να υποβάλει μια νέα πρόταση μέχρι το 2016 εισάγοντας πραγματικές συνθήκες δοκιμών στην πραγματική οδήγηση που θα οδηγούν στο να συνάδουν αυτές οι εκπομπές ρήπων. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιανκόφσκα, κυρία Πίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σήμερα συζητάμε την θέσπιση της νέας διαδικασία δοκιμών για τις εκπομπές για τα οχήματα, τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργαζόμασταν όπως ξέρετε επ' αυτού επί μακρόν χρονικό διάστημα, αλλά βεβαίως χρειάζονται εφαρμοστικοί κανονισμοί επιγόντως και διατάξεις θα εστιαστώ λοιπόν στη συζήτησή μου, στην αναφορά μου, στον αντίκτυπο που έχουν οι ληφθήσεις αποφάσεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι αξιόπιστες οι δοκιμές στα εργαστήρια. Οι πραγματικές εκπομπές από, το από τις είναι 400 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο όσον αφορά τα ζωτούχα. Τέσσερις με πέντε φορές υψηλότερο το ποσό αυτό από το νόμιμο όριο των αυτοκινήτων που έχουμε καθορίσει τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό έχουμε προτείνει αλλαγές όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και βέβαια ήταν απαιτητικό ο στόχο αυτό. Καταλήξαμε σε μοναδική λύση, η οποία πετυχαίνει το σκοπό τη κατά την άποψή μα. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, ή θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, θα θεσπίσουμε δοκιμέ για τι εκπομπέ σε πραγματικά οχήματα, πραγματικού δρόμου, υπό κανονικέ συνθήκε οδήγηση. Οι λύσει μα θα αλλάξουν το σύστημα μετρήσεω εξ ολοκλήρου. Δεν θα είναι πλέον εφικτό κανείς να κλέψει όσον αφορά τις δοκιμές εκπομπών. Κατέληξαν τα κράτη-μέλη σε συμβιβασμό. Στα 168 μιλιγκράμμ ε, ανά χιλιόμετρο θα περιοριστούν οι εκπομπές μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο του χρόνου και μέχρι τον Ιανουάριο 2020 θα μειωθούν οι εκπομπές περαιτέρω σε 120 ε, μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Θα γνωρίζετε ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο φιλόδοξες. Επανειλημμένα είπα ότι ήθελα αυστηρότερους παράγοντες συμμορφώσεως. Δεν μπορούσαμε όμως να πείσουμε τα κράτη-μέλη. όλα αυτά, και το υπογραμμίζω αυτό, θεωρώ ότι η συμφωνία αποτελεί ουσιαστική πρόοδο, διότι οι εκπομπές αζωτούχων των δυσλοκινητήρων μειώνονται κατά το ίμιση. Και πιέζουμε και την αυτοκινητοβιομηχανία να επιταχύνει τις προσπάθειες ούτως ώστε τα αυτοκίνητα να γίνουν καθαρότερα και να σεβαστούν τους κοινού ε, περιβαλλοντικούς μας στόχους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τους νέους κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν τάχιστα. Γι' αυτό ζητούμε και τη σύμφωνη γνώμη σε αφορά την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση πραγματικών ε, δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω σα είπα όμω, δεν θα σταματήσουμε εδώ οι πραγματικές αυτές οι δοκιμές, οι πραγματικές συνθήκες είναι ένα κομμάτι της δέσμης μέτρων. Θέλουμε να μειώσουν τις κομπές των αζωτούχων όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν μάλιστα οι τεχνικές εξελίξεις που μας επιτρέψουν θέλουν τα αυτοκίνητα να φτάσουν στα 80 ε, μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο. Γι' αυτό η πρόταση νομικού ε, περιεχομένου προτείνει ετήσια αναθεώρηση, ρήτρα ετησία αναθεωρήσεω. Δηλαδή, από το 2020 και μετά, τα όρια αυτά θα μπορούν να προσαρμόζονται αν βελτιωθεί η αναλόγω η τεχνολογία. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί ε, την τεχνολογία όσον αφορά τι μετρήσει, ούτω ώστε να γίνονται μετρήσει υπό πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και αν βελτιωθεί η τεχνολογία μετρήσεων και επιτρέπει ακριβέστερη μέτρηση εκπομπών το 2020 και μετά, θα υπάρχει νομική δυνατότητα τα όρια να μειωθούν έτσι περαιτέρω, να φτάσουμε στα 80 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε το έργο αυτό από το τέλος του ενεστώτος έτους. Και είναι δυνατό να γίνει αυτό ε, εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου μέχρι το τέλος του έτους. Επειδή οι κατασκευαστές σχεδιάζουν τα οχήματά τους πολύ πριν την παραγωγή τους, ούτω ώστε τα οχήματα στους δρόμους σε πέντε χρόνια ήδη τώρα σχεδιάζονται. Γι' αυτό η ύπαρξη της ρήτρα περιετησίας αναθεωρήσεως παρέχει ασφάλεια δικαίου και δίνει κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία να σχεδιάζει τα οχήματά της με πολύ χαμηλότερες εκπομπές από ό,τι τα παρόντα όρια. Στρέφομαι τώρα στο υπόλοιπο πακέτο. Κατά τη διάρκεια του έτου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τρίτο ρυθμιστικό πλαίσιο για πραγματικέ δοκιμέ στι συνθήκε οδήγηση για βελτίωση τη διαφάνεια. Ποια είναι η ιδέα ότι οι παράγοντε συμμορφώσεως κάθε οχήματο θα πρέπει να φαίνονται στο πιστοποιητικό συμμορφώσεως. Ο καταναλωτής θα έχει πλήρη επίγνωση των εκπομπών ε, του αυτοκινήτου του ή αυτοκινήτου της. Έτσι δε περαιτέρω, δεσμεύομαι να βελτιώσω το σύστημα ε, εγκρίσεω και θα βελτιωθεί η ανεξαρτησία των φορέων ε, έγκρισης και θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Οι νέοι κανόνες θα θεσπίζουν και θα ενισχύουν το σύστημα που υπάρχει και θα ε, γίνει αυστηρότερο το σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει και να σχολιάζει τα συλλογικά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Το σύστημα ανταλλαγή των πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολή του νόμου των κρατών μελών θα ενισχυθεί. Είδαμε επίση ότι τα κράτη-μέλη δεν αντιδρούν συντονισμένα. Γι' αυτό προτίθομαι να υποχρεώσω τα κράτη-μέλη να διενεργήσουν έρευνε αγορά και να ελέγχουν αυτοκίνητα που διατίθενται στην αγορά. Η ποιότητα και ανεξαρτησία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνε για την έγκριση των οχημάτων θα είναι κάτι που θα πρέπει να ενισχυθεί. Άρα χρειάζονται περισσότερες δοκιμές ποιοτικέ, καλύτερη συνεργασία και καλύτερα εργαλεία για την επιβολή των διατάξεων. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας όσον αφορά τις εγκρίσεις τύπου, το σχετικό σύστημα και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το συμφωνήσαμε άλλωστε όταν το συζητήσαμε προηγουμένω. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κατεπηγόντω νέου κανόνε για τι εγκρίσει τύπου και τι δοκιμέ εκπομπών. Και κάτι εξίσου σημαντικό. Να πω καλά λόγια για τι προτάσει που γίνονται. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαπραγματεύονται κάποιε αναθεωρώσει τη νομοθεσία Euro 5 και Euro 5 και Euro 6 που αφορά την θέσπιση κανόνων για τον έλεγχο εκπομπών υπό πραγματικέ συνθήκε. Θα δοθούν κατησοδότηση εξουσία εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητούνται αυτέ, Θέλουμε ομαλή και ταχύ εφαρμογή ε, τη νέα διαδικασία στο μέλλον. Θα συνεργαστούμε μαζί σα και με το Συμβούλιο βέβαια. Θέλουμε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. Θέλουμε να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και είμαστε αποφασισμένοι να σεβαστούμε τη διαθεσμική ισορροπία. Γνωρίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό αυτό και για σας αξιότιμα μέλη. Ελπίζω ότι οι δεσμεύσεις μου είναι σαφέστατες για σας. Θέλω να είμαι συνεπής και πλήρης στην προσέγγιση μου. Θα ζητήσω αποφασιστική κίνηση κατά των αυτοκινητοβιομηχανιών αν δεν συμμορφωθούν. Το νέο πλαίσιο θα αποκαταστήσει την αποτελεσματικότητα του νομικού μας συστήματος. Έτσι θα προστατεύουμε και τους καταναλωτές και το περιβάλλον και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ξεκινάμε τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μπέλετ είναι ο πρώτος ομιλητής. Uh, ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό περί του οποίου πρόκειται είναι τα οξύδια αζότου, οι εκπομπές ε, οξυδίων αζότου και πρέπει τάχιστα να μειωθούν αυτές οι εκπομπές και το Euro 6, Euro 6 για τα οχήματα diesel που τετραπλάσιο όγκο αζωτούχων ε, εκπέμπει σήμερα πρέπει τάχιστα να μειωθούν τα επίπεδα εκπομπών ρήπων οξυδίων του αζότου και τα, οι δοκιμές πραγματικές συνθήκες οι νέες δοκιμασίες είναι αναγκαίες και συμφωνούμε επ' αυτού. Μόνο που χάσαμε χρόνο, σπαταλήσαμε χρόνο δυστυχώς. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θα υποβληθεί μια νομική πρόταση από πλευρά σας. Είναι αναγκαίο το δυνατόν γοργότερα να υποβληθεί. Η εθνική έλεγχη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να είναι ανεξάρτητη στο χαρακτήρα τους και πρέπει η έλεγχη αυτή να είναι αποτελεσματική. Αναφέρομαι στις διατάξεις ε, και στις νομικές πράξεις και η συζήτηση από αυτού εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει άμεσα να ληφθεί υπόψη και θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όταν πρόκειται κατεξουσιοδότης για κατεξουσιοδότηση πράξης ε, να προχωρήσουμε με τον πιο ευφυή τρόπο για τις ε, ευφυείς τεχνολογίες. Δεν θα αναμείνουν οι αυτοβιομηχανίες της αντιδράσεις ε, αν καθυστερήσουμε. Ήδη εξετάζουν τις νέες τεχνολογίες στην εφαρμογή τους. Κύριε Μπέλετ, ο κύριος Σάνι έχει σηκώσει γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε? ο κύριος Ζάνη λοιπόν. Να θέσετε το ερώτημά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον συνάδελφο που δέχεται την παρέμβαση. Ιδιαίτερα θέλω να ζητήσω να υπάρξουν αυστηροί κανόνες και να προσαρμοστούμε, να τηρήσουμε αυτούς τους αυστηρούς κανόνες Πώς όμως θα γίνουν όλα αυτά. Να μην είναι υπερβολικά αυστηροί αυτοί οι κανονισμοί. Και όταν βλέπουμε ότι η καθυστέρηση να δράσουμε. Κύριε συνάδελφε, αγαπητέ συνάδελφε, θα πρέπει να πω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι να συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα σε σχέση με αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, τα σκάνδαλα τα οποία είδαμε και βιώσαμε και να συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση. Σημαντικό είναι τα οξύδια του αζότου να μειωθούν. Έχουμε μια εξεταστική επιτροπή που θα δει και και θα διαπιστώσει τι πήγε στραβά, τι δεν έγινε σωστά. Και πιθανότατα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι δοκιμασίες έγκρισης τύπων, τύπων οχημάτων θα πρέπει να αυστηροποιηθούν με ανεξάρτητους ελέγχους. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που πήγαν στραβά. Έχουμε μια εξεταστική επιτροπή και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε και να δούμε πώς το δυνατόν γοργότερα θα μειωθούν τα οξύδια του αζότου. Είναι σημαντικό για τη δημόσια υγεία για όλους μας. Κύριε Μπέλετ, είστε πολύ δημοφιλή με τις Ο κύριος Στά, λοιπόν θέλει να το κουβεντιάσει αυτό. Δέχεστε. Καλώ, κύριε Στα, ορίστε. Σα ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία πρόεδρε. Κύριε Μπέλετ, ουσιαστικά θα ήθελα να ρωτήσω Πώς εκπροσωπείται η ομάδα σας και όταν σε δύο, μήνες, σε δύο εβδομάδες θα ψηφίσουμε για αυτή την ένσταση, ένσταση θα υπερψηφίσετε τα μελήματα και τις ανησυχίες μας υπέρ της δημόσιας υγείας ώστε να εξευρεθεί μια πραγματική λύση και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση. Αν δεν υπερψηφίσετε όμως θα σημαίνει αυτό ότι τις ισχύουσες διατάξεις τις παλαιότερες θα τις υποστηρίζετε που είναι υπερβολικές και υπερβολικές εκπομπές ε, ρήπων. Πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα σας λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ κύριε Στάς για την ερώτησή σας. Η δική μας ομάδα φυσικά θα υπερψηφίσει υπέρ της δημόσιας ε, υγείας. Η κυρία Επίτροπος ανέφερε ότι τα σημερινά οχήματα τετραπλάσιες ποσότητες ρήπων ε, εκπέμπουν από ό,τι κατά το παρελθόν. Γι' αυτό πρέπει πραγματικά να δράσουμε και μετά από δύο, δυόμιση έτη να υπάρξει σημαντική μείωση κατά το ίμιση των εκπομπών και μετά από δυόμιση περαιτέρω έτη να ξαναμειωθούν οι εκπομπές οξυδίων του αζότου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση η οποία έχει οξυνθεί και με τα οχήματα αυτά και τους ελέγχους να προχωρήσουμε. Η απόφαση θα πρέπει να είναι κατά το ίμιση μείωση και περαιτέρω μείωση μετά. Ευχαριστώ. Κυρία Βαν Μπρέντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στους προλαλήσαντες. Δεν χρειάζεται να επαναληφθούν όλα τα επιχείρηματα εκ νέου πραγματικά θα πρέπει οι δοκιμασίες αυτές οι δοκιμές να γίνονται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η ομάδα μας όμως υπεψήφισε μία αναβολή ώστε να υπάρξει κάποιο περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να βελτιώσει τα πράγματα με την πρότασή της σωστά επιχειρήματα και σωστές ε, είναι οι προθέσεις αλλά χρειάζονται πιο φιλόδοξες ε, δράσεις. Δεν είναι αποδεκτό ότι κάποια τεχνική επιτροπή θα λαμβάνει τελεσίδικα αποφάσεις τι θα γίνει με την κατηγορία Euro 6, Euro 6 που αποφασίσαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ επανεξετάστε το και βελτιώστε την πρότασή σας σε σχέση με τον συντελεστή συμμόρφωσης 1 ένα, μόνο ένα. Μόνο έτσι θα, θα συνάδουν με τις δημοκρατικές προοπτικές ε, οι προτάσεις σας. Να υποβάλλετε λοιπόν μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Ευχαριστώ. κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό που θέλουμε είναι καλύτερη ποιότητα του σφαιρικού αέρα. Θέλουμε τεθεί τέρμα στι εγκρίσει τύπου μέσω εργαστηρίου και θέλουμε πραγματικέ συνθήκε να επικρατούν στι δοκιμέ το ταχύτερο δυνατόν. Βέβαια υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειε προς συμφωνία, αλλά η θεμελιώδη συμφωνία βρίσκεται επιτάπητος από την 28 Οκτωβρίου στη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει πραγματική αλλαγή. Μέχρι το 2020 θα έχουμε εγγυημένο παράγοντα 1,5 συμμόρφωσης, παράγοντα συμμόρφωσης. Κάποια οχήματα που είναι στους δρόμους τώρα εκπέμπουν 5 με 6 φορές παραπάνω το όριο των 80 mg. Πώς μπορείτε να απορρίψετε τη δυνατότητα να περιορίσετε και να φτάσουμε στα 120 mg; Ο λαός της Ευρώπης, που έχει ο κόσμος που έχει αμπευστικά προβλήματα λόγω μόλις στην Ευρώπη, το αξίζει αυτό. Θέλουμε ένα παράγοντα συμμόρφωσης 1 και θέλουμε να δεσμευτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κατημέρια. Θα το πετύχουμε αυτό με συγκεκριμένε ημερομηνία. Υποστήριξη του στόχου ε, απλώς μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσει και καθυστερήσει έτη και μήνε δεν θέλουμε. Δεν θα βελτιωθεί η υγεία δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Α αρπάξουμε την ευκαιρία. Α καθίσουμε στο τραπέζι. Α συμφωνήσουμε. Ο... Θα πρέπει να συμφωνήσουν με τον παράγοντα συμμόρφωση σε ένα τα κάτι μέλη. Να μην υπάρχει μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τελικά όλοι να κάνουμε προσπάθεια να συνοηθούμε. Ο κύριο Γκερμπράντι έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις παρεμβάσεις σας. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θέλω το εξή να τονίσω. Και δεν πρέπει αυτό να το αγνοήσουμε φυσικά στη συνέχεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες στην Ευρώπη αυτό το θέμα. Επιθυμούν να είναι καθαρός και υγιής ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναπνέουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και να μην απειλούνται από τους ρήπους των οχημάτων. Και κυρία Επίτροπε, η δική σας Επιτροπή λέει ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη νομοθετική δράση, better regulation, καλύτερη νομοθετική ε, δραστηριοποίηση. Ωστόσο, αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν θα πετύχετε αυτό το στόχο, δεν θα υπάρξουν μελέτες επιπτώσεων και κανείς ε, δεν θα είναι υπεύθυνο στη δράση που αναλαμβάνει. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο ε, να δούμε ότι απουσιάζει πλήρως ε, στη απόψηνή μας συζήτηση. Και αυτό θα πρέπει στα κράτη-μέλη να ασκήσουμε επικρίσεις εις βάρος τους, μια και δεν διασφαλίζεται η, καθαρή, η ποιότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα. Και θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό του καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Να ερωτήσω την Επίτροπο, πώς θα μπορέσουν οι πολίτες μας στις πόλεις της Ευρώπης να επιβιώσουν όταν αντιμετωπίζουν έναν ατμοσφαιρικό αέρα που έχει μολυνθεί από τις εκπομπές ρήπων των οχημάτων. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας λοιπόν για τη διασφάλιση της ε, υγείας των πολιτών μας. Λοιπόν, θα έπρεπε ε, ήδη οι οριακές τιμές ε, να ισχύουν για το 2016 και βλέπουμε ότι έχουν υπερ, έχουμε υπερβεί αυτές τις τιμές. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διασφαλιστεί καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας υπέρ των πολιτών μας. Το 2015 στην Ολλανδία υπήρξαν πολλές διακηρύξεις και ακούστηκε ότι το software αυτό που ε, χρησιμοποιήθηκε ήταν παραπλανητικό, εξαπάτησε και όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει επιτέλους τα κράτη-μέλη να προβληματιστούν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική στο μέλλον. Η παραπλανητική αυτή πολιτική απάτης πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτέλους. Η κυρία είναι η επόμενη που έχει το λόγο λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένας Ευρωπαίος στους δύο ζει στις πόλεις. Και εκεί τα μεταφορικά μέσα ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δημιουργεί 430.000 πρώιμους θανάτους το χρόνο. 940 δι σε κόστος όσον αφορά την υγεία. Όταν λοιπόν μιλάμε για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς. Πώς είναι δυνατόν να μην ελέγχουμε τις εκπομπές των οξυδίων του αζότου. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 80 μιλιγκράμμ που έχουμε καθορίσει σαν όριο, ανά χιλιόμετρο. Πρέπει να τηρήσουμε τα 80 και όχι να πηγαίνουμε ε, από 168 και να κατέβουμε σε 120 κλπ. Χρειαζόμαστε ένα όριο περιοριστικό. Δεν θα πρέπει να θέτουμε σε να εμποδίζουμε και τους μηχανισμούς ε, ε, που προβλέπει ο κανονισμός. Θα πρέπει να επαναξεταστεί ο κανονισμός που διέπει αυτά τα στοιχεία. Ελπίζω ότι θα είμαστε θέση ε, από τώρα και σε 10 χρόνια να πούμε ότι καταφέραμε να ελέγξουμε τις εκπομπές των οξυδίων του αζότου και θα εξοικονομήσουν και πολλά χρήματα έτσι. Διότι όπως σας είπα αυτό αντιπροσωπεύει πολλά όσον αφορά τις δαπάνες του τομέα της υγείας. Δισεκατομμύρια ευρώ αντιπροσωπεύει. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε μια νέα πρόταση πολύ πιο φιλόδοξη για να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Ο κύριος Αϊκχάουτ έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Mike, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο που εξε... την Επίτροπο που εξήγησε άλλη μια φορά το πρόβλημα. Ε, απογοητεύομαι λίγο γιατί ε, δεν ε, άκουσα για μία ακόμα φορά ποια πιθανή αλλαγή μπορεί να προέρχεται από την πρόταση. Και αυτό που άκουσα από εσά, κύριε Επίτροπε, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγή. Τα, τα κράτη-μέλη άκουσα ότι όλα τα οχήματα μπορούν να εκπέμψουν μέχρι 168 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2019 και αναφερθήκατε μόνο στην ημερομηνία για τα νέα μοντέλα. Αλλά πρέπει να αναφερθούμε σε όλα τα μοντέλα. Και υπάρχει και ο, ο παράγον ε, συμμόρφωση 1,5 που σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε φτάσουμε στα 120 ξεκινώντας μόνο το 2021 παρότι ήδη από το 2007 εμείς ως συνομοθέτες αποφασίσαμε ότι θα πρέπει το 2014 να πάει στα 80. Αυτό κάναμε ως συνομοθέτες. Αυτό που γίνεται τώρα στην τεχνική συνεδρίαση είναι να λέμε ότι αυτό αυτό, το νούμερο μπορεί να πάει στα 120 μέχρι το 2021. Άρα, ακόμα κι αν είναι κανείς στα χέρια της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν μπορεί να αποδεχτεί. Σε μια τεχνική επιτροπή προσαρμόζουμε, διορθώνουμε αυτό που αποφασίσαμε ως συνομοθέτες. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τώρα πλέον μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ καλύτερα. Σήμερα τα, στα φλαμανδικά νέα με ένα αυτοκίνητο, με μια απλή διόρθωση πήγε από 750 στα 200 σε μία μέρα και τώρα συμφωνείτε ότι υπάρχει χρόνος μέχρι το 2021 για να για να υποβαθμίσουν μια πρόταση που θα έπρεπε να είχε ε, που άλλαξε η ημερομηνία. Οι σοσιαλδημοκράτες ρωτούν, θα υπάρχει νέα πρόταση για τους παράγοντες συμμόρφωσης, ναι ή όχι. Και θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και η Ιταλική Αντιπροσωπεία και το κίνημα των Πενταστερών υποστηρίζουν αυτή την ένσταση, διότι αντιμετωπίζουμε πραγματικά μια ένα ξεγέλασμα. Προτείνεται το πακέτο αυτό σαν ε, μεγάλο βήμα προόδου, σαν ένα μέτρο άκρος φιλόδοξο και μοναδικό στον κόσμο. Κρίμα που εκ των πραγμάτων, πώς μπορεί να είναι κάτι φιλόδοξο και μεγάλο βήμα προόδου κάτι τέτοιο, ένα πακέτο το οποίο θα επιτρέψει παρόλα αυτά στα οχήματα να μολύνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τα όρια τα οποία επιτρέπονται. Είναι γεγονό και πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι οι επιχειρήσει τη αυτοκινητοβιομηχανία είχαν 7 χρόνια στη διάθεσή του να μπορέσουν να προετοιμαστούν και να τακτοποιηθούν και να σεβαστούν τα όρια ε, υπό πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Αυτό δυστυχώ όμω δεν έγινε και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια. Απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά να προτείνει το ταχύτερο δυνατόν ένα μέτρο, επαρκέ μέτρο και σοβαρό που θα προστατεύει την υγεία των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνάνο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα πολύ δυσάρεστο δίλημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια καλή ιδέα να ε, μειώσει τις ε, απαιτήσει ε, ε, των ελαφρών, εκπομπών των ελαφρών οχημάτων, ε, είτε λάβουμε υπόψη μας την υπόθεση Volkswagen όχι, πρέπει να, να, να, πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή αυτοκίνητο βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλη ανεργία και για μία ακόμα φορά η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη Για μία ακόμα φορά κινείται με τον αγαπημένο της τρόπο παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, διαφάνεια και ανάληψη ευθύνη. Το κοινοβούλιο αυτό θα έπρεπε να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει την υπερβολική γραφειοκρατία. Αλλά βεβαίω ο οικονομικό πόλεμο έχει ξεκινήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε και γι' αυτό θα αντιδράσουμε σε αυτή την αντίδραση. Ο συνάδελφο Λίζε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Αληθεύει κάθε χρόνο αποβιώνουν 400.000 ε, πολίτες πρόωρα λόγω της ε, μόλυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Και πολλές φορές ε, οι ευθύνες βρίσκονται ακριβώς στο θέμα της τήρησης αυτών των τιμών για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Γι' αυτό θα πρέπει στην γη να συνεχίσουμε την προσπάθεια μείωση των ρήπων. Φυσικά σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν και τα οχήματα. Θέλουμε μια λύση για το real drive emissions, τις πραγματικές εκπομπές ε, ρήπων υπό πραγματικές συνθήκες και να δούμε τι μπορεί να γίνει και να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Όμως το θέμα του τι συμβαίνει εδώ δεν είναι τόσο απλό να βρούμε τις απαντήσεις του. Μια πλειοψηφία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είπε ότι η πρόταση δεν είναι αρκετά αυστηρή, γι' αυτό την απορρίπτουμε. Και σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη υπάρχουν και λόγοι θετική για να γίνει κάτι τέτοιο επειδή η Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια αυστηρότερες ε, τιμές ε, είχε αρχικά προτείνει Ωστόσο όμως μπορούμε να πούμε ναι ή όχι, να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε και γνωρίζω από προσπάθειες που γίνονται από πολιτικούς που εμπλέκονται και στο Συμβούλιο με την απόρριψη της πρότασης δεν θα υπάρξει μια πιο αποτελεσματική ρύθμιση ή πιο αυστηρές τιμές. Γι' αυτό εμείς από το ΕΛΚ είμαστε υπέρ ενός συμβιβασμού που θα βοηθήσει τους πολίτες για την υγεία τους και δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας στο σχεδιασμό από την άλλη πλευρά σε σχέση με την αυστηροποίηση και την αδειοδότηση οχημάτων. Ελπίζω τις επόμενες δύο εβδομάδε θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντεγκρούτε, έχετε το λόγο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι γερμανικές πόλεις έχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την τήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Τι να πούμε στους δημάρχους ε, των πόλεων μας με αυτή την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε συντελεστές επιδίνωσης που απορρέουν από την Ευρω 6 και καταλήγουμε στην Ευρω 5 ρύθμιση. Τι μπορούμε να αναμένουμε αν υπάρχει ένα συμβιβασμό ως προοπτική για τον οποίο εργαζόμαστε και ελπίζουμε να υπάρξει ένα τέτοιο συμβιβασμό και οι συντελεστές ε, ε, συμμόρφωσης για την επιδείνωση τι μπορούν να συνεισφέρουν. Τι θα πούμε στους δημάρχους. 20 χρόνια θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία από το 2007 στο 2027 ή ποια θα είναι η καταληκτική ημερομηνία τελικά Πώς το αντιμετωπίζετε. Βλέπετε τον κίνδυνο ίσως για την τήρηση των οριακών τιμών για τον ατμοσφαιρικό αέρα να αντιμετωπιστεί η προοπτική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Επιτροπής. Βλέπετε μια τέτοια προοπτική ή όχι και είσαστε άνετοι. Και όσον ε, αφορά το θέμα που είναι τόσο σημαντικό, πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια τώρα να συζητήσουμε. Όμως το Συμβούλιο απουσιάζει και αυτό είναι ντροπή, έσχος. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρέτσελ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μείωση των οξυδίων του αζότου σίγουρα είναι ένας στόχος που μας συνενώνει όλους υπέρ αυτού του στόχου. Και αυτό το εξέφρασαν όλοι οι προλαλήσαντες απόψε. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε σήμερα πάρα πολλές επικρίσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας που ακούστηκαν. Όμως κυρίες και κύριοι δεν φταίει η αυτοκινητοβιομηχανία για τους κανονισμούς αυτούς, αυτούς ως έχουν σήμερα για την έγκριση τύπων οχημάτων που πειραματικά εκπονούν κάποιοι με δοκιμές. Δεν είναι απάτη της αυτοκινητοβιομηχανίας αυτή όπως ακούστηκε από διάφορους προλαλήσαντες είναι απλά η ανικανότητα των πολιτικών να καταλήξουν σε δοκιμασίες, σε τεστ τα οποία θα βρίσκονται κοντά στην πραγματική λειτουργία και συνθήκες λειτουργίας των οχημάτων. Γι' αυτό αν μπορέσουμε επ' αυτού να συμφωνήσουμε στο μέλλον κάτι θα έχουμε καταφέρει. Και όπως ανέφερε ο συνάδελφος Μπέλετ, ανέφερε την ευφυή αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο κανένας δεν έκανε λόγο για την ΕΦΗ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή απουσιάζει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τόρβαλτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι απλό και να το σκεφτούμε αυτό που θα θέσω σαν ερώτημα. Σε μια νομοθετική διαδικασία τι γίνεται όταν υπονομεύεται το νομοθέτημα από εκείνους που δεν είναι αξιωματούχοι, δεν υπονομεύονται οι δημοκρατικές αρχές. Θα πρέπει να ο καθένας αλληλοκατηγορείται σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα αυτό, κάτι πρέπει να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε τα μάτια έναντι τεράστιων των εκπομπών και τώρα βιάζεται να θα σπίσει μέτρα. Η Volkswagen διέπραξε απάτες. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε περισσότερα και πρόσεχε περισσότερο θα μπορούσε να είχε προστατεύσει την εφαρμογή των ποδιαγραφών της. Έχει ευθύνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς να λέει ότι είναι πολύ οργά να κινηθούμε και ότι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Ντελή. Η απόφαση που ελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο είναι σκανδαλώδης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, τα κράτη-μέλη επέτρεπαν στην αυτοκινομήχανία να ρηπαίνει. Θα μπορούν πλέον να ξεπερνάνε τα κατά 110% το... μέχρι το 2020 και 50% μετά. Σκανδαλώδες και θα πρέ, μας λένε ότι είναι και παράνομο η υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή είναι μια παραβίαση ε, κατάφορη όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι συνομοθέτης. Οι κανόνες για την προστασία της υγείας των πολιτών δεν γίνονται σεβαστές. Και είναι κοινοφελή μέτρα. Εμείς δεν εξυπηρετούμε τα λόμπι της αυτοκινητομηχανίας. Αντί να είμαστε συνένοχοι τη βιομηχανία, το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξουν το στατόπεδο των πολιτών, των καταναλωτών και του πλανήτη. Αυτή η απόφαση σκανδαλώδη θα πρέπει να απορριφθεί από τον επόμενο μήνα. Καλό τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν το ίδιο και να επιληθούν του θέματος. Θα πρέπει να θεσπίσουν πραγματικούς ελέγχους ε, ανεξάρτητη αδειοδότηση και έγκριση θα πρέπει να γίνεται. Γίνονται πραγματικέ δοκιμέ σε πραγματικέ συνθήκε και αυτό θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Γιάουκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, το σκάνδαλο που που ξέσπασε στην γερμανική αυτοκινοβιομηχανία τον περασμένο Σεπτέμβριο αποκαλύπτει ανησυχητική ανισορροπία ανάμεσα στα πρότυπα των ρήπων και την πραγματικότητα του κλάδου. Συμφωνώ ότι σε αυτό το ψήφισμα πρέπει να ασχοληθούμε με, το, με, την επίδραση στην υγεία και δεύτερον τα πρότυπα. Επιπλέον προστίθεται ένα επιπλέον ε, όριο σε, μια, ε, έναν κλάδο που διώκεται. Και όλα αυτά με τη φροντίδα της οικολογικής, της, οικολογικής, της πολιτικής της οικολογίας πρέπει να επιβεβαιώνουμε ότι η μείωση των, εκπομπών, των ρήπων θα γίνει με τη μείωση των διεθνών ροών, ένα είδος από παγκοσμιοποίησης που κανείς ούτε καν οι, πολιτικοί οικολόγοι δεν θέλουν να αναφέρουν εδώ. Και ε, σε αυτό ε, πρέπει να, κάτι να κάνουμε. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για τη μείωση των ρήπων στην ατμόσφαιρα μεταξύ αυτών και των διοξιδίων του αζότου. Οι μέχρι τώρα πρακτικές ε, των δοκιμών στα εργαστήρια δεν ήταν ε, διαφανείς, είναι απαράδεκτες γιατί οι συμπολίτε μας πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν. Γι' αυτό η οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για όλους τους αυτοκινητοβιομηχανίες ε, είναι, σημαντικό, ε, είναι σημαντική. Όμως ε, υπάρχει μια αντίρρηση εδώ γιατί αν ψηφίσουμε την, την πρόταση της Κομισιόν θα καθυστερήσει σημαντικά αυτές τις καλύτερες δοκιμές που είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις παλαιότερε που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Άρα είναι πιο υπεύθυνο για το περιβάλλον και για την αυτοκινητοβιομηχανία να ε, μην στείλουμε σε ελληνικέ να στείλουμε σε ελληνικές καλένδες το κείμενο. Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας αλλά και να διατηρήσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι λοιπόν, αν εγκρίνουμε αυτή την αντίρρηση θα ε, θέσουμε ε, ε, εμπόδια ενώ το status quo θα είναι το ξεκίνημα μιας λύσης. Θα μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο πολιτικοί στο μέλλον για τις ε, εκπομπές των, της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά αυτό όμως πρέπει να γίνει πλαισιώνοντας ε, τον κλάδο στην μεταβατική αυτή περίοδο είναι θέμα εμπιστοσύνης που πρέπει να, να υπάρχει στους συμπολίτες μας και για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας που αποτελεί σημαντικό. Περιμένουμε η Κομισιόν να πάρει ισχυρά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση για να ε, γίνονται καλύτεροι έλεγχοι στις δοκιμές αυτές. Διακοπή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ντάλη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε.

η οποία αναφέρει ότι βαίνουν λέει, όλα καλώς και θα μπορούν να τηρούνται αυτές οι τιμές. Ωστόσο η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά είναι πολιτικού χαρακτήρα απόφαση. Ο ρόλος των πολιτικών είναι να διασφαλίζουν τους πολίτες τους ε, σε συγκεκριμένα ζητήματα και θέλω να ερωτήσω να απευθύνω ερώτηση προς τους ε, Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και την πίεση αυτή που οδηγεί σε διπλάσιες εκπομπές ρήπων μέχρι το 2020 και τι θα γίνει σε σχέση με την πολιτική που θέλουμε να ακολουθηθεί μέχρι το 2020. Δεν είναι η χρονική στιγμή να υπαναχωρήσουμε έναντι των πιέσεων των λομπιστών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και θέλω να ρωτήσω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και ποιες εγγυήσεις δίνονται σήμερα για μια θετική προοπτική. Ο κ. Κράμερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέραμε εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν απάτες, ότι ψέματα, ψεύδι διαχέονται και αυτό αναφέρθηκε και σε σχέση με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Δεν έγινε όμως τίποτα. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας. Η τεχνολογία υπάρχει, υφίσταται. Είναι θέμα κονδυλίων, χρημάτων τα οποία θα απαιτηθούν. Και σε σχέση με τα οχήματα diesel που επιδοτούνται σε πολλές χώρες, παρόλα αυτά συνέβη αυτό. Στη Γερμανία 18 σεντ λιγότερα πληρώνουν οι καταναλωτές για ένα λίτρο diesel σε σχέση με ένα λίτρο βενζίνης και κάτω από 90 σεντ σήμερα. Αυτά όμως μπορεί να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πορευτούμε. Ο έντιμος πολίτης ε, δεν πρέπει να είναι ο χαζός, ο βλάκας, ο οποίος θα εξαπατάται και θα πληρώνει και περισσότερα. Δεν πρέπει αυτοί να τιμωρηθούν όσοι τηρούσαν τα όρια και τις τιμέ Πρέπει να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι εξαπάτησαν και διέδωσαν ψεύδι. Γι' αυτό λοιπόν οι τιμές που έχουν εγκριθεί πρέπει να οδηγήσουν στο να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο κ. Σβάμπ, για 1,5 λεπτό. Ο κ. Σβάμπ, κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν με σαφήνεια να τονίσω ότι κανείς την μείωση των οξυδίων του αζότου δεν την αμφισβήτησε. Το αντίθετο, όλοι συμφωνούμε. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί στη στοχοθέτησή μας. Όμως εδώ δεν πρόκειται για αποζημιώσεις ε, για τους πολίτες που επλήγησαν, παρότι και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πρέπει να δούμε αν ε, οι νομικές πράξεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτονται ή εγκρίνονται από εμάς. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν τις απορρίψουμε όπως προτείνετε εσείς, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι το περιβάλλον θα εξασφαλιστεί στην ποιότητά του. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσετε γιατί θέλετε να υπομισθούμε αυτό τον κίνδυνο και να διακυβευθεί η υπόθεση αυτή. Μπορεί να μην είναι η πιο ικανοποιητική κατάσταση αυτή, όμως είναι ίσως το καλύτερο βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Και σκεφτείτε και προβληματιστείτε αν μπορείτε να συμπορευτείτε μαζί μας. Το ότι δεν είναι απλό αυτό το κατανοώ. Δεν θέλουμε οι έντιμοι να πληγούν και να υποστούν κυρώσεις. Και υπάρχουν μια σειρά ολόκληρη δυνατοτήτων για βελτιώσεις που διανοίγονται ενώπιόν μας. Όμως συνάδελφοι, όχι στη διαδικασία διαδικασία αδειοδότησης των οχημάτων ΙΧ. Σε άλλους τομείς ε, πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει για να προσαρμοστούν τα πράγματα, να συνεργαστούν καλύτερα τα κράτη-μέλη και να μην, να μην διαπιστώνουμε στο τέλος ότι δεν τηρούνται όσα αναφέρθηκαν. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε μάχη από πλευρά τη ομάδα μας. Πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταλήξει στην ε, αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ε, για την έγκριση νομικών πράξεων και για τη στοχοθέτηση σε στόχους που μας συνενώνουν. Παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η, η απόφαση της Επιτροπής που συζητάμε σήμερα πήρε την απόφαση την ίδια μέρα που το Κοινοβούλιο έθεσε ε, πολύ φιλόδοξους στόχους για τις εθνικές εκπομπές. Αυτό μας παρουσιάστηκε ως τεχνική αλλαγή, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πολιτική. Ό,τι είναι βρώμικο σκοτώνει. Τώρα μόλις έχουμε συνειδητοποιήσει το εύρος του πόσο ο βρώμικος αέρας σκοτώνει τους πολίτες αλλά από το 2006 γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και τις πραγματικές εκπομπές. Ήδη η Επιτροπή το αναγνώρισε το 2011. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κατάσταση όπου 10 σχεδόν χρόνια μετά τις αρχικές εκθέσεις θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια καθυστέρηση των πολύ απαραίτητων πραγματικών δοκιμών και των προτύπων που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπή. Επίτροπε. Δεν μπορούμε να, γίνονται, να λαμβάνονται αποφάσεις τελευταία στιγμή πριν αποκλειστέ πόρτες. Πρέπει να, να ακολουθήσουμε έναν συνεπή δρόμο που θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα και αυτό έχει σχέση και με την λογοδοσία αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριο Βάντεν Κάμπ. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ από πλευράς μου πιστεύω ότι απόψε δεν πρέπει να αποκρύψουμε ένα πράγμα. Το 2015 ήταν ένα πολύ αρνητικό έτος για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία οι καταναλωτές, οι αρχές έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν σαφείς έντιμες πληροφορίες για την καθαρότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το δίλημα ε, στα, τα επόμενα έτη. Οι συνάδελφοι, για παράδειγμα, όπως ο κύριος Λίζε, ανέφεραν πράγματα. Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει ένα ε, αυστηροποιημένο πλαίσιο, ε, στοχοθέτηση η οποία θα τηρηθεί με δοκιμασίες υπό πραγματικές συνθήκες, real driving tests. Και εδώ πρέπει πραγματικά οι ε, διεθνείς ε, υπηρεσίες και φορείς να δραστηριοποιηθούν. Επίτροπε μπορείτε να μας δώσετε σαφείς ε, προοπτικές το τι μπορεί να γίνει με συγκεκριμένα χειροπιαστά βήματα που θα ακολουθηθούν. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι χάνουν σιγά σιγά την υπομονή τους. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και να παραμείνουμε στην πραγματικότητα. Τι μπορεί να γίνει πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι να παρεκκλίνουμε. Πρέπει να δούμε και την ε, σύνοδο για την προστασία του κλίματος στο Παρίσι. Ε, πρέπει να δούμε γιατί όλα αυτά ε, σε σχέση με τις ΗΠΑ αποκαλύφθηκαν και όχι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σέρτουκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε θα έλεγα Πιστεύω η μπάλα είναι στο δικό σας γήπεδο, στην Επιτροπή. Πρέπει να το πούμε. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη ως εκτελεστικό σκέλος για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και το πρόβλημα αυτό πρέπει να τύχει δίκαια λύσης τώρα. Είναι αδιαμφισβήτητο αυτά από τα τους τεχνικούς οργανισμούς και φορείς απορρέων και σε σχέση με την πρότασή σας ε, δεν ήταν αποδεκτά. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτό που θέλουμε να γνωρίζουμε από εσά είναι οι απαντήσεις σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, την αρχή των real driving emissions θα την ακολουθήσετε την αρχή αυτή των πραγματικών δοκιμών νέου. Η δεύτερη ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι υπηρεσίες της επί ολόκληρα χρόνια τις επισημάνσεις των εθνικών φορέων για αυτά τα θέματα τις αγνόησαν. Διότι αυτό πρέπει να απαντηθεί για να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρντίνη έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω εγώ ότι η συζήτηση που διεξάγεται στην αίθουσα αυτή μας βρίσκει όλους ενωμένους. Προς μια κατεύθυνση κινούμεθα και προσπαθούμε να κινηθούμε επί μακρό, να βελτιώσουμε δηλαδή την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Επ' αυτού δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Επί δεκαετίε η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη βελτιώθηκε πάρα πολύ. Καλό αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, διότι δεν αρκεί αυτό. Σίγουρα. Θα πρέπει όμως να συνδέσουμε την οικολογία με την οικονομία. Αυτό το έλεγε ένας ενδιαφέρον αρθρογράφος σε μια τελική εφημερίδα. Η οικολογία, το κίνημα του οικολογικό φαίνεται να πουλά την υγεία στους πολίτες, όμως την πραγματικότητα κάνει κακό και στην υγεία των πολιτών. Γιατί αν εμείς εδώ ακολουθήσουμε τη λογική εκείνων που σήμερα ισχυρίζονται ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι του περιβάλλοντος, οι καλύτεροι προσπιστέ τη ποιότητα του νοσφαιρικού αέρα θα βρεθούμε με τεράστια αντίφαση. Θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ αυτή τη ένσταση και θα βρεθούμε με μια διολίστηση διετία όσον αφορά τι διαπραγματεύσει και τελικά δεν θα επιφέρουμε τη βελτίωση τη ποιότητα του νοσφαιρικού αέρα που αν ψηφίσουμε ναι, αντιθέτω θα την έχουμε αμέσω και θα εφαρμοστούν αμέσω τα μέτρα. Σήμερα εδώ βλέπετε συζητούμε αν θα ψηφίσουμε περαιτέρω σημαντική μείωση όσον αφορά τι εκπομπέ σωματιδίων και οξυδίων του αζότου. Δύο από τα, τις χειρότερες αιτίες ε, για ασθένειες και ε, θανάτους. Θα πρέπει με ειλικρίνεια και σαφήνεια να το αντιμετωπίσουμε κατάματα και να υπερψηφίσουμε και θα πρέπει να, να βοηθήσουμε τουλάχιστον τη βιομηχανία να βρει την τεχνολογία η οποία τελικά θα είναι καλύτερη και θα πετυχαίνει τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παουλούτσι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ε, κυρία Πρόεδρε, μέσω ημών με ύψιλον θα ήθελα να απευθυνθώ στο Συμβούλιο και εκφράζω τη θλίψη μου και τη διαμαρτυρία μου διότι απουσιάζει το Συμβούλιο από αυτή τη σημαντική συζήτηση. Χρειάζεται μεγαλύτερο σεβασμό από πλευρά του Συμβουλίου όσον αφορά τι εργασίε του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα πια είναι σαφέ ότι οι μετρήσει που γίνονται στο εργαστήριο όσον αφορά τι εκπομπέ οξυδίου του από τι κινητήρε δίζελ των αυτοκινήτων είναι τρει ή τέσσερι φορέ χαμηλότερε από τι πραγματικέ συνθήκε στις συνθήκες οδήγησης. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια όσον αφορά τη ρήπανση ατμοσφαιρικού αέρα. Επί σειρά ετών ε, διαμαρτύρεται κοινή γνώμη. Και τους λέμε ψέματα. Είχαμε μετά το σκάνδαλο της Volkswagen. Ευπρόσδεκτο λοιπόν αυτό ότι θα θέλουμε να έχουμε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Ζητούσαμε επί σειρά ετών Κανεί δεν θέλει να στραγγαλίσει την βιομηχανία, αλλά θέλουμε σοβαρότητα στον αντιμετώπιση του προβλήματο. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε τα 80 ε, μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο σαν όριο. Πώ γίνεται να δεχόμαστε λοιπόν αυτό το όριο από το 2021 μετά από 15 χρόνια να φτάσει στα 120. Όχι. Δεν αληθεύει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η υγεία στις πόλεις μας χρειάζεται πιο απαραίτητε επεμβάσεις. Εμείς θα πρέπει να μην θελοτυφλούμε και να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, το θάμο στην άμμο. Ευχαριστώ η κυρία Αγιούζο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι θέλουμε καλύτερη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καλύτερο περιβάλλον. Είναι αυτονόητο. Να απορρίψουμε όμως αυτόν τον κανονισμό είναι ακριβώς το αντίθετο αν απορριφθεί αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να δούμε τι θα μπορεί να γίνει για την βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις μας παρακολύοντας σε σχέση με τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Αυτό που έχουμε στο τραπέζι είναι οι Ευρω 5 και Ευρω 6 ρυθμίσεις για την ρύθμιση των εκπομπών ρήπων των οχημάτων υπό πειραματικές συνθήκες. Υπό πραγματικές συνθήκες πολλαπλασιάζονται όμως αυτές οι εκπομπές ρήπων Κάνουμε λόγο λοιπόν για ένα συντελεστή συμμόρφωσης τεσσάρων, τετραπλάσιο δηλαδή, σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές ε, ρήπων. Και ο συντελεστής ρύθμισης ε, ε, είναι 2,1 για το 2007 και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα δεν μπορούν να μετρηθούν σε πραγματικές συνθήκες οι εκπομπές ρήπων με μεγαλύτερη σοβαρότητα χρειαζόμαστε ε, καλύτερες ε, προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να τις βρούμε και να δράσουμε ώστε να υπάρχει κατά 100% ε, σεβασ, ε, Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν απορριφθεί αυτός ο κανονισμός θα καθυστερήσουμε τρι, δύο ή τρία χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και πρέπει να δούμε ότι το περιβάλλον εδώ δεν ε, εξυπηρετείται. Εδώ έχουμε της ε, δράσης μιας επιτροπής ε, εξέτασης ε, που πρέπει να μας κάνει να δράσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Η κυρία έχει το λόγο το να κάνουμε αυτό που λέμε και να λέμε αυτό που κάνουμε είναι ένας συνεπής κώδης συμπεριφορής. Μετά τον κώδικα 21 και τους φιλόδοξους ε, στόχους, το πώς να δεχτούμε αυτά που ζητάει η Κομισιόν που επιτρέπει στο πρότυπο, επιστρέφει στο πρότυπο Euro 6. Οι, γαλλικές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί στην πραγματικότητα, στην πράξη, οι εκπομπές ε, είναι πολύ πιο είναι διαφορετικές από ότι στο εργαστήριο ε, και χρειάζομαστε όλο και πιο ε, εντυπωσιακά αυτοκίνητα. Δεν ζούμε στα, ε, στο εργαστήριο. Είναι πολύ καλό να αναγνωρίζονται οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, αλλά κυρίως να μην μειώσουμε τις απαιτήσει. Μήπως αποφασίστηκε η αύξηση του τορίου ταχύτητας. Βεβαίως και όχι το Γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να ε, ασχοληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί με το θέμα. Πρέπει να επέλθει καλύτερο συμβιβασμός για τον, για τον σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων. Τον Φεβρουάριο έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι και εσείς θα, ε, να δείξετε ότι και εσείς θα κάνετε αυτό που πρέπει. Ο κύριος Κάμπους για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να βρούμε το ερώτημα το εξής που πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις. Αυτή η κατάσταση μας οδηγεί στο να προχωρήσουμε ή καθυστερεί τα προγράμματα για τη μείωση εκπομπών στην Ευρώπη. Είναι καλό το ότι έχει δεσμευθεί να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια δέσμη μέτρων σαφέστερη και πιο μετρήσιμη. Γιατί θα πρέπει να παραμείνουμε στην πραγματικότητα για να έχουμε τα εχέγγυα, να καταλήξουμε σε στόχους που θυμούμε. μείωση των εκπομπών ρήπων των οξυδίων του αζότου αποτελεσματικά. Πρέπει να επαγρυπνούμε λοιπόν στη στάση μας όσον αφορά τις διατάξεις ε, επανεξέτασης. Πρέπει να επαγρυπνούμε εναντί των βιομηχανιών. Όμως το γράμμα του νόμου δεν μπορεί να προχωρήσει πιο μπροστά από την τεχνολογία. Διότι διαφορετικά θα αποτύχουμε και η αποτυχία θα αφορά την υγεία και τις θέσεις εργασίας. Στα καταλανικά ελπίζουμε ότι το νέο έτος θα φέρει υγεία και απασχόληση και εργασία. Θέλουμε όμως να υπάρχει μια Ευρώπη η οποία θα προχωρήσει έτσι και δεν θα είναι Ευρώπη άνεργη. Ρεαλιστικά πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρώπη ώστε να είμαστε πιο πράσινοι στη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργία πρόσθετης αξίας. Ευρώπη που θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις ε, που αναλήφθηκαν στην Σύνοδο για την Προστασία του Κλίματος στο Παρίσι. Αν καθυστερήσουμε και υιοθετηθεί η πρόταση ε, απόρριψης ε, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα είμαστε, είμαστε λοιπόν κατά της ένστασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαντεμός έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να γίνονται δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Οι μετρήσεις σε εργαστήριο τελικά δεν είναι πετυχημένες. Είναι απαράδεκτο αυτή η αλλαγή να χρησιμοποιείται όμως για να επιτρέπονται μεγαλύτερα επίπεδα εκπομπών οξυδίων του αζότου. Και είναι κάτι αντιπαραγωγικό αυτό. Κάποιοι από εμά βλέπουμε την ομοθεσία, τη δέσμη μέτρων για τον σφαιρικό αέρα που έχουν σαν στόχο τη μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε ότι αρκετέ χιλιάδε ε, συμπολιτών μα ε, πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω προβλημάτων ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα. Εμεί έχουμε ένσταση κατά τη προτάσεω αυτή, διότι οδηγεί σε περισσότερη ρήπανση. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Σας παρακαλώ να ετοιμάστε μια πρόταση που θα οδηγεί σε αποτελεσματικό σύστημα δοκιμών χωρίς να υπάρχουν κενά και χωρίς πολλούς συμβιβασμούς όσον αφορά την υγεία των πολιτών μας. Και τώρα ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. Κυρία Επίτροπε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αρκετά τυχοδιοκτική αυτή η συζήτηση που διεξάγουμε συμφωνήσαμε για οριακές τιμές. Όλοι γνώριζαν ότι πειραματικά μετρώνται αυτές οι τιμές και όχι στις υποπραγματικές συνθήκες. Μετά υπήρχε το, υπήρξε το σκάνδαλο της Volkswagen και εργαζόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνιμα για να βρει μια ε, διαδικασία ε, για την... Ε, τον καθορισμό των τιμών που θα είναι πιο αποτελεσματική. Και άμεσα υπήρξε αντίδραση και μια ρεαλιστική πρόταση που υποβλήθηκε. Όμως δεν επενέθηκε η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κατηγορήθηκε και αυτό είναι αντιστροφή των όρων. Τώρα έχουμε διαδικασία υπό πραγματικές συνθήκες, όλοι το επιθυμούσαν, το έχουμε υπό τιμές που είναι ε, εφικτές ε, για αυτές ε, τις δοκιμασίες και γοργά οι υπεύθυνοι για την υγεία των πολιτών αν επιδεινωθεί η κατάσταση είναι εκείνοι οι οποίοι θα εγκρίνουν αυτή την ένσταση για να μιλάμε ξεκάθαρα εκείνοι οι οποίοι την πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου την απορρίπτουν για το ότι θα υπάρχει επί χρόνια επιδεινωμένη κατάσταση στους δρόμους μας αυτή είναι η πραγματικότητα εκείνοι που θα συνεργαστούν και θα διασφαλίσουν να υπάρξει ταχύτερα μια ρύθμιση για την βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όχι βέβαια ονειρική και ιδανική, αλλά καλύτερη και βήμα προς βήμα δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει βελτίωση στη συνέχεια. Λοιπόν, τι θα αποφασίσετε, υπέρ της βελτίωση ή υπέρ της επιδείνωσης. Thank Σας ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στη δικασία Κατστιάη. Πρώτος, πρώτη κυρία Σόιτε Μπίρικ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα στους συναδέλφους για τη συνεργασία, για την αναζήτηση μιας λύσης. Η ερώτηση είναι αν η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να αποδείξουν ότι αυτή η ρύθμιση κατά 105 ή 110% θα είναι νομικά κάτι το οποίο θα μπορεί να ε, υπερασπιστούμε. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ τις ε, νομικές διατάξεις ε, που βλέπουμε ότι παρακάμπτονται. Αύξηση και υπέρβαση σημειώνεται. Υπάρχουν παρεκκλήσεις λοιπόν με τις ίδιες τις μετρήσεις και τις συσκευές μετρήσεων. Και βλέπουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εδώ δεν είναι δυνατό να οδηγήσει στην τήρηση αυτών των τιμών ακόμα και όσον αφορά τους καταλήτες. Αναφέρθηκε ότι πρόσθετοι λέει καταλήτες μπορούν να εξοπλίζονται, να τοποθετούνται στα οχήματα και η Volkswagen και όλα ε, από πλευράς ε, τεχνικής προοπτικής ανέφερε κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αυτοκινητοβιομηχανίας να εξευρεθεί μια λύση. Η αυτοκινητοβιομηχανία λέει ότι θέλει να είναι υπόδειγμα. Ε, όμως αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Να σε υπενθυμίσω μόνο ένα λεπτό μπορεί να μιλάει ο καθένας στο ΚΑΤΣΤΙΑ. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Παρακαλώ τηρήστε το χρόνο. Επόμενος ο μιλητής ο κ. Μπλάνκο Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι εκθέσεις ε, για ε, την εξαπάτηση σε σχέση με τις εκπομπές ρήπων θέτει την αυτοκινητοβιομηχανία εν ώψη μιας ε, περίπλοκης και δεινής κατάστασης. Και σε σχέση με την ίδια την Ισπανία όπου αεξατώνται 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ως υπεύθυνοι για τον δημόσιο βίο υποχρεούμεθα να λάβουμε συνετά, συνετές αποφάσεις που θα διευκολύνουν την λειτουργία αυτού του τομέα, θα προστατεύουν τους εργαζόμενους, θα δίνουν εγγυήσεις στους καταναλωτές που αγοράζουν αυτά τα οχήματα και θα είμαστε αποτελεσματικοί για τις εκπομπές ρήπων ώστε να μειώνονται αυτές σταδιακά υπέρ του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι στις πραγματικές συνθήκες οι δοκιμασίες είναι υποχρέωση. Υποχρέωση όχι μόνο η νομική αλλά κατεπίγουσα ανάγκη για τους πολίτες. Και ζητούμε αυτό το κατεπήγον να μπορέσει να συνάδει με την μείωση των εκπομπών ρήπων από πλευρά τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εκτιμώ ότι υπάρχει εδώ ομοφωνία. Θα ήθελα όμως να πω ότι λυπάμαι για τη θέση του Συμβουλίου. Δεν είναι έντιμη στάση το απέναντι στο Κοινοβούλιο με το, από το γεγονός ότι δεν παρίσταται σήμερα. Παρά τα αυτά, εργαστηριακές δοκιμές δεν ήταν ρεαλιστικέ. Παρά, παρόλα τα αυτά έγιν, γίνονταν. Υποτίθεται ότι η, η, ήταν σε συνθήκε πραγματικού κόσμου. Αλλά βεβαίω υπήρχαν αμφιβολίες. Εκτιμώ αυτά που είπε σήμερα η Επιτροπή. Η πρόταση όσων είναι κατά της πρότασής της θα είναι αντιπαραγωγική. Φυσικά είμαι υπέρ πιο καθαρού αέρα, όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για και να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πράγματι η παρατήρηση που έχω να κάνω πρώτη είναι η απουσία του Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες στη συζήτηση. Ε, οι συνάδελφοί μου έχουν δίκιο όταν λένε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και αυτό όχι μόνο στον τομέα των αυτοκινήτων. Εγώ είμαι πολύ διστακτική, διότι αν απορρίψουμε αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και τις μετρήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα ε, είναι πολύ ευρύ το πλαίσιο γενικά και αόριστο. Δεν ξέρω αν η αναβολή που θα προκύψει θα είναι εποφελής για τους ε, καταναλωτές. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Γι' αυτό Λοιπόν, εγώ διστάζω για αυτή την προσέγγιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά όταν είναι να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε για το σχέδιο του κανονισμού. Πάντα το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμασμάκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευτυχώς που υπάρχουν ε, οι δημοσιογράφοι που κάνουν έρευνες. Ιδάλλως θα είχαμε κι άλλη απάτη με την δίθεν αναβαθμισμένη διαδικασία για την ε, εκ των υστέρων εγκατάσταση των, των διαφόρων μοντέλων. Ένας φλαμανδός ε, δημοσιογράφος ε, έχει κάνει έρευνα ε, πρέπει ως καταναλωτές να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με σοβαρότητα. Αν εγώ πρέπει να επιλέξω ε, ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που είναι πιο ισχυρό ή έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ένα ταχύτερο αυτοκίνητο είναι καλύτερο ε, για τα παιδιά μου, θα επιλέξω αυτό που είναι καλύτερο για την υγεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία. Είμαστε εμείς το Κοινοβούλιο. Το οφείλουμε στους πολίτες να δείξουμε αυτού του είδους τη φιλοδοξία. Ευχαριστώ. Θα σταματήσουμε εδώ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά άλλα αιτήματα, αλλά δεν έχουμε αρκετό χώρο να ε, ανταποκριθούμε σε όλα. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ. Οπότε τώρα δίνω το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος στον κύριο Γιάβορ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Επίτροπε, από τη σημερινή συζήτηση καταλήγω ότι σήμερα από επαγγελματική σκοπιά συμφωνούμε ότι ο παράγων συμμόρφωσης που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι ρεαλιστικός, είναι γελίος. Ακόμα και η Επιτροπή το θεωρεί ανεπαρκή για την επίτευξη των στόχων μας. Έγινε πολλή συζήτηση για καθυστέρηση, αλλά είμαστε ειλικρινεί. Ο κανονισμός θα τεθεί ενισχύ το 2019. Έχουμε λοιπόν χρόνο να τον βελτιώσουμε και να ασχοληθούμε κάπως περισσότερο με έναν με τη βελτίωσή του για την δημιουργία ενός κανονισμού που προστατεύει το περιβάλλον και τους πολίτες. Και πραγματικά αυτή η προσέγγιση είτε αυτό είτε το συμφωνείτε είτε δεν, δεν έχετε τίποτα απέναντι στο Κοινοβούλιο δεν ε, θεωρώ ότι είναι δημοκρατική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό το, λοιπόν θέλω να σας, υποστηρίξω, να, να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτή την αντίρρηση και να κάνετε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να καθίσουν και πάλι στο τραπέζι για τη βελτίωση του κανονισμού. Αντί να είσαστε ρεαλιστές, να είσαστε θαραλέοι και παραγωγικοί Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Και τώρα η Επίτροπος Μπιενκόφσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις και τις θέσεις σας. Έχω... Σέβομαι τις ανησυχίες σας και τις κατανοώ θα επιστρέψω στα πιο βασικά ερωτήματα. Και πάλι όμως θα υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή δεν αγνόησε οποιαδήποτε προηγούμενη ένδειξη, ούτε το 2006 όταν δουλεύαμε για την πρόταση του Euro 5-6 για, να, για τη μείωση των εκπομπών. Αυτό όμως αφορούσε εργαστηριακές δοκιμές και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Το 2011 και το 2012 είχαμε το GRC και κανένας άλλος που είπε για πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόβλημα με τις εκπομπές. Τώρα, με τη θετική ψήφο και πάλι αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας, με τη θετική ψήφο πρέπει να σταματήσει, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούμε να προτείνουμε οτιδήποτε νέο όσον αφορά τους παράγοντες συμμόρφωσης. Γιατί? Επειδή καταρχήν τα κράτη-μέλη δεν θα αλλάξουν την άποψή τους. Δεύτερον, θα καθυστερήσει πάρα πολύ την όλη διαδικασία αυτό. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αν δεν υπάρχουν κανόνες το 2017, θα διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή θα παραμείνει η κατάσταση με εκπομπές 4-5 φορές υψηλότερες στην πραγματική ζωή και θα έχουμε πολύ περισσότερη μόλυνση. Η απόρριψη θα σημαίνει ότι το 2017 δεν θα υπάρχουν κανόνες, οπότε θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες μας. Γιατί έχουμε τώρα 500 μιλιγκράμμ ε, εκπομπών διοξιδίου του αζότου ε, ανά χιλιόμετρο και δεν κάναμε τίποτε όμως ε, μπορεί να υπάρξει συνένεση ελπίζω και υπάρχει ενδεχομένως ένας πιθανός τρόπος να προχωρήσουμε χωρίς νέες προτάσεις και παράγοντες συμμόρφωσης η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να κάνει μία δήλωση στην ψηφοφορία της ολομιλίας τον επόμενο μήνα περιγράφοντας ε, τη λύση που προτείνουμε σήμερα ειλικρινά θέλω να ενεργοποιηθεί ο, η ρήτρα ετήσιας αναθεώρησης για τον επόμενο παράγοντα συμμόρφωση των επόμενων έτος που σημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό ε, με την ε, χρήση του παράγοντα αυτού και δεύτερον θα βελτιωθούν οι ε, έρευνες για την ε, πραγματική οδήγηση. Αυτό αποτελεί δεσμευσή μου. Ελπίζω ότι αυτό θα επιτρέψει τουλάχιστον σε κάποιους από εσά να ψηφίσετε υπέρ των προτάσεων για τις ε, ε, εκπομπές την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να πω ότι έχουμε πρόταση αυτή την πρώτη ψηφίσματος πέρα στη συζητήσεως. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο. Και τώρα επιθυμίσω κάτι από τον κανονισμό, σας παρακαλώ. Κάτι διαδικαστικό μάλλον. Κύριε Γκερμπράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε την Επίτροπο. Ανέλαβε υποχρεώσει για το μέλλον. Η απόφαση που ελήφθη όμως αυτά τα μέτρα είναι απόφαση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς δεσμεύσει από το Συμβούλιο. Οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κενέ, θα έλεγα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα αυτό στο Συμβούλιο να του ζητήσετε απάντηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις που να λάβατε, ούτως ώστε να λάβουμε γραπτή απάντηση από τα απόν ε, Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέμπραντι, Δεν ήταν διαδικαστικό αυτό που θέσατε, έτσι δεν είναι. Ε, Πρόκειτο περί παρεμβάσεως πολιτικής φύσεως. Επόμενο σημείο λοιπόν. Έχουμε έκθεση της Επιτροπής ε, Πολιτισμού για το ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολυμορφίας της πολιτισμικής και πρόθεση των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα δώσω το λόγο, περιμένετε, να ψάξω να βρω το όνομα.